Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Να σας δώσω τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας. Εψήφισαν 725 691 είναι οι έγκυρες 346 είναι η απόλυτη πλειοψηφία. Η κυρία Φορέντσα έλαβε 42. Η κυρία Λάμπερτ 51 ψήφους. Ο κύριος Πιτέλα 200 ψήφους. Ο κύριος Ρεμπέγκα 45. Η κυρία Στέβενς 66 ψήφους. Ο κύριος Ταγιάννη 287 ψήφους. Διαπιστώνω ότι κανείς υποψήφιος, ούτε υποψήφια δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, οπότε θα προχωρήσουμε αναγκαστικά σε τρίτο γύρο εκλογής Προέδρου. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θεωρώ ότι οι υποψηφιότητες του δευτέρου γύρου διατηρούνται και για τον τρίτο γύρο της εκλογής Προέδρου. Μέχρι στιγμής Έχω την κυρία Φορέντσα, την κυρία Λάμπερ, τον κύριο Πιτέλα, τον κύριο Ρεμπέγκα, την κυρία Στέβενς και τον κύριο Ταγιάννη ως υποψηφίους. Αλλά και στον τρίτο γύρο αυτό μπορούν να κατατεθούν και νέες υποψηφιότητες πριν τον τρίτο γύρο. Γι' αυτό ορίζω προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιότητων ή αλλαγές σε σχέση με τις υποψηφιότητες ε, ε, στην πέμπτη απογευματινή. Αυτέ οι υποψηφιότητε θα πρέπει να κατατεθούν στον πρόεδρο που διευθύνει τη ε, συνεδρίαση στο γραφείο της Προεδρίας για νέα υποψηφιότητα. Θα πρέπει όλα αυτά να υποβληθούν στον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Προθεσμία λοιπόν 5 το απόγευμα και 5.30 θα συνεδριάσει και πάλι ολομέλεια και μέχρι τότε διακόπτεται.